Ας ξεκινήσουμε. Έχετε όλη την κάρτα ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε Ευχαριστώ.

questa. Αν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι.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 με την ε, τροποποίηση του κανονισμού 1234-2007 του Συμβουλίου ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ για την ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του γερμανικού μονοπωλίου αλκοόλης. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε συνέχεια της συζήτησης στην Επιτροπή μας με τους συναδέλφους και τους προσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, εξασφαλίσαμε την μεταβατική και όχι στρεβλωτική φύση του στην εσωτερική αγορά αυτή της έκθεση, η οποία παρατείνει το μονοπόλιο αλκοόλης της Γερμανία, επομένω υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η θέση αυτή ε, βασίζεται με θετική στήριξη και από το Συμβούλιο. Έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε σε συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση θεωρώ αναγκαίο να υποβάλω μια τροπολογία για την μέγιστη διαφάνεια στην σταδιακή κατάργηση. Ε, υποχρέωση αναφοράς στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Κάμια άλλη τροπολογία δεν έχει υποβληθεί, επομένως προτείνω να περάσουμε άμεσα στην ψηφοφορία. Ψηφοφορία διανατάσεως της χειρός. Καταρχήν, Ψηφίζουμε για την τροπολογία του εισηγητή. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την νομοθετική πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τέλος ψηφίζουμε για την πρόταση, την νομοθετική πρόταση και το ψήφισμα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. Ωραία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Εγώ δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ας περάσουμε γρήγορα γρήγορα στην ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος για τις μέλισσες, για τη μελισσοκομεία. Έχουμε διάφορες τροπολογίες. Ευτυχώς όμως, χάρη στην εργασία της κυρίας Λούλινγκ, την οποία ευχαριστώ, ε, υπήρξαν πολλές συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Ας, χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα. Παρακαλώ βάλετε την ε, κάρτα σας και προετοιμαστείτε. Αν έχετε ετοιμαστεί, ας ξεκινήσουμε. Έχετε την... τον κατάλογο της ψηφοφορίας. Ωραία, ας ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ας ξεκινήσουμε με τη συμβιβαστική πρόταση 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία συμβιβαστική 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνατε οι δύο. Συμβιβαστική πρόταση 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 3. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ζήτησε το λόγο για την παράγραφο 45 ο κύριος Λαβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα απλώς να εξηγήσω το περιεχόμενο της 45 για να είναι σαφές το νόημα της ψηφοφορίας. Ε, τα προγράμματα γίνονται με βάση την ε, εκτίμηση ε, των αριθμών των κρατών μελών. Η τροπολογία θέλει τα προγράμματα να γίνονται με βάση τα προγράμματα καταγραφής των μελισσών, όχι σε εκτιμήσεις, για να αυξηθεί έτσι η διαφάνεια στη χρήση των κοινοτικών πόρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λαβία. Ας ψηφίσουμε τη 45. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 45. Προχωρούμε. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 5. Αρχίζει. Πέρας της ψηφοφορίας για την 5 εγκρίνεται. Ας περάσουμε στην 6. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 6. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 7. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε τώρα την ε, τροπολογία 60. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 60. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 63. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 63. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Ψηφοφορία για την 64. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίπτεται και αυτή. Ας περάσουμε τώρα στη συμβιβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία για την 8. Πέρας της ψηφοφορίας για την 8 εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για την τροπολογία 68. Άρχεται η ψηφοφορία για την 68. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Η κυρία Γέγκλ έχει ζητήσει τον λόγο. Ελίζαμπεθ. Αποσύρω αυτή την τροπολογία διότι το περιεχόμενο περιλαμβάνεται σε άλλες. Καλώς. Δεν ψηφίζουμε λοιπόν για την 69. Αποσύρθηκε 69, δεν την ψηφίζουμε. Τροπολογία 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραστε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 72. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 74. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 74. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας για την 74 απορρίπτεται. Τώρα, περνάμε στην συμβιβαστική τροπολογία 10. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 10. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται η συμβιβαστική τροπολογία 10. Περνούμε στην συμβιβαστική τροπολογία 9. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την ενεά. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται η συμβιβαστική τροπολογία 9. Τροπολογία 84. Άρχεται η ψηφοφορία Ταραμπέλα μπάτζι. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφοφορία για την 85. 85. Άρχεται η ψηφοφορία. 85. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίας απορρίπτεται. Περνούμε τώρα στην 87. Ντάντζιλα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία για την 87 απορρίπτεται. 88. Αρχίζει η ψηφοφορία. 88. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 89. Αρχίζει η ψηφοφορία. Της κυρίας Γέγκαλ. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 90. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ενημερώθηκα ότι υπήρχε μια πλεονάζουσα ψήφος από το Λαϊκό Κόμμα. Παρακαλώ να γίνει έλεγχος. Πάντοτε παραπάνω ο οπαδοί του Λαϊκού Τροπολογία 91 των Ράιμερς και Λούλινγκ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 91. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 93. Σιλβέστρης. Αρχίζει. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 93. 95. Τον Ταραμπέλα Ταμπάτζη. Άρχεται η ψηφοφορία για την 95. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 96. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 96. Πέρας της ψηφοφορίας για την 96. Απορρίπτεται. Πάλι έχουμε μια πλεονάζουσα ψήφο από το ΕΛΚ. Κάποιος παραπάνω ψηφίζει. Προσοχή. Ο Ζωσέ Μποβέ προτείνει αντίπεινα προτείνει να τη δώσουμε στους πράσινους αυτή την ψήφο. Ας ανοίξουμε την ε, ψηφοφορία. Α, καταπίπτει η 97 του Νικουλέσκου. Περνάμε στην 98. 98 Νικουλέσκου. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 98. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ας περάσουμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Πρώτη τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Αρχίζει η ψηφοφορία για τη 2. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συνεχίζουμε με τις ιδεολογικές σκέψεις. Τρία. Γκαρσία, Περές και άλλοι. Ψηφίσατε όλοι για την τρία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στην συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 11. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 11. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 7 του Χάρκιν. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 7. Α, συγγνώμη, ε, συμπεριλαμβανόταν. Οπότε περνάμε στη συμβιβαστική τροπολογία 12. Σε δύο χωριστά μέρη. Πρώτο μέρος. Αρχίζει η ψηφοφορία για το πρώτο μέρος. Πέρας της ψηφοφορίας για το πρώτο μέρος της συμβιβαστικής τροπολογίας 12 εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε τώρα το δεύτερο τμήμα της 12. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τώρα περνούμε στην τροπολογία 9. Όχι. Όχι, περνούμε στην τροπολογία 13. Ρέιμερς και άλλων. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τροπολογία 13. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14. Συμβιβαστική τροπολογία 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 13. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 23. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέραστη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25 των Γκαρσία Πέρες και άλλων. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε τη συμβιβαστική πρόταση 15. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τελική τροπολογία 32. 32 άρχεται η ψηφοφορία για την 32. Πέρας της ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Και τώρα ο τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ σε όλους. Τώρα θα περάσουμε απευθείας στην Ολομέλεια. Μετά από αυτή την ψηφοφορία θα πάει η έκθεση στην Ολομέλεια. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στο 11ο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έτοιμη Ντατσάνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα της έκθεσης Σάρμπου, αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισυτιστικής ασφάλειας, είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, στρατηγικής φύσεως. Η εκθετική ανάπτυξη των της κατανάλωσης σε πολλές περιοχές του κόσμου ε, ενέχει το κίνδυνο να περάσουμε σε ένα σενάριο όπου τα τρόφιμα θα γίνουν ένα σπάνιο και ακριβό αγαθό. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις του Ηνωμένων Εθνών, το 2005 θα φτάσουμε στο ένα δισεκατομμύριο. Και το θέμα της διατροφής θα αποκτήσει πολύ μεγάλη σημασία θα φτάσουμε σε επάρκεια τροφίμων του 70%. Όχι μόνο η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα των τροφίμων θα αλλάξει δραστικά. Η μεγαλύτερη, ε, το μεγαλύτερο εισόδημα του πληθυσμού θα δημιουργήσει σε πολλές υποκαταστάσεις στο καλάθι της νοικοκυράς. Και γι' αυτό τη στιγμή αυτή που συζητούμε το ρόλο της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, η έκθεση, της, ε, ε, η έκθεση Σάρμπου θα αποκτήσει, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δίνω λοιπόν το λόγο στην εισηγήτρια και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι χαίρομαι πολύ διότι έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά με τους συναδέλφους. I know it, is it's also Romanian, so it shouldn't be a problem. Oh. No, no. Ναι. Δεν είναι πρόβλημα της διερμανίας. Παρακαλώ, σβήστε το μικρόφωνο καταρχήν. Ένα λεπτό παρακαλώ να λυθεί ένα πρόβλημα με τον μεταφραστικό εξοπλισμό. Yes. Είναι εντάξει αν χρησιμοποιήσω αυτό το μικρόφωνο. Okay, Ας δούμε τώρα αν λειτουργήσει το σύστημα. Siamo? Έτοιμοι. Ας δοκιμάσουμε. Λοιπόν, ξαναξεκινάω. Ε, ε, θα επαναλάβω και την εισαγωγή. Ήθελα να σας πω από την αρχή ότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με τους συναδέλφους και τους ευχαριστώ για τις ιδέες τις οποίες παρουσίασαν και που με βοήθησαν να παρουσιάσω αυτή την έκθεση για το μέλλον της Ευρώπης. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να τονίσω τις βασικές ιδέες και θα ακούσω με τα χαράς και την δικιά σας γνώμη. Και βεβαίως θα γίνει και ένας διάλογος επί αυτού. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι η επισητιστική ε, ασφάλεια είναι η βάση της νέας γεωργικής πολιτικής μετά το 2013. Η γεωργία είναι ένα τομέα κλειδί για την ασφάλεια, τη διατροφική ασφάλεια και για την καταπολέμηση της φτώχειας και την ανάπτυξη των λαών και γι' αυτό τώρα ε, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ε, υπάρχουν μεγάλες αλλαγές κλιματολογικές, μεγάλες προκλήσεις, ε, σημαντικές κλιματολογικές αλλαγές, λιγότεροι πόροι και πολύ ψηλές τιμές ενεργείας και γι' αυτό θα έπρεπε όλοι να λάβουν υπόψη αυτές τις παραμέτρους παραμέτρους για, που επηρεάζουν τη διατροφική ασφάλεια να προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν τις διακοιμάνσεις των τιμών για να εξασφαλίσουν ε, μια ομαλή προμήθεια τροφίμων. Χαιρετίζουμε τα ε, τα μέσα τα οποία μας πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο κανονισμού και την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πολλά παραπάνω. Ε, παραδείγματος χάρη να καταπολεμήσει και να περιορίσει την κερδοσκοπία με μέτρα τα οποία θα μειώσουν τις διακοιμάνσεις των τριμών ε, να ε, επεξεργαστεί περισσότερο τα χρηματοοικονομικά μέσα για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και να επιτρέψει να συμμετάσχουν σε αυτή την αγορά περισσότεροι. Ε, επιπλέον όσον αφορά τις διακοιμάνσεις των τιμών βλέπουμε ότι είναι όλο και πιο ευαίσθητη η προμήθεια τροφίμων υπάρχουν μεγαλύτερες κρηματολογικές στρατηγικές διακυμάνσεις και ε, όπως σας είπα αυτή τη στιγμή έχουμε αποθέματα μόνο 12 εβδομάδων. Άρα η ΟΗΕ θα πρέπει να επιβλέπει αυτά τα αποθέματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει μία ηγετική θέση σε αυτό το σύστημα καθότι η διατροφή είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου και δεν πρέπει απλώς να μιλάμε αφηρημένα αλλά να προτείνουμε ουσιαστικά μέτρα. Οι αλλαγές τις οποίες πρότεινα θα πρέπει να λάβουν χώρα στα πλαίσια μιας ε, γενικότερης ε, κοινής ε, γεωργικής πολιτικής η οποία πρέπει να είναι πιο ισορροπημένη, να υπάρχει καλύτερη ισορροπία να μην υπάρχουν κράτη των οποίων η θέση απειλείται. Ε, επίσης θα πρέπει να υπάρξουν προτεραιότητες ε, στην γεωργία, να διατηρήσουμε την στήριξη στην παραδοσιακή γεωργία και ε, να εξασφαλίσουμε μία ποικιλότητα των τροφίμων διότι βλέπουμε ότι ε, θα μειωθούν σύντομα ή γεωργοί. Έχουμε 4,5 εκατομμύρια τα γεωργούς οι οποίοι σύντομα θα συνταξιοδοτηθούν άρα χρειαζόμαστε να ανακαινήσουμε το επάγγελμα και να τους βοηθήσουμε με πιστώσεις. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένας προϋπολογισμός ώστε όλοι να μπορέσουν να υποφεληθούν και όλες οι διαδικασίες σε αυτήν την έκθεση ε, έχουν εξεταστεί από την σκοπιά της ε, νέας ε, κοινή γεωργικής πολιτικής η οποία θα πρέπει να είναι πολύ πιο ισοσκελισμένη και ελπίζω ότι θα έχουμε έναν πιο επικοδομητικό διάλογο με νέες ιδέες. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε αμέσως τη συζήτηση. Ας ξεκινήσουμε από τον κύριο Χάιουαρθ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την εισηγήτρια και να χαιρετήσω την ε, έκθεση αυτή, γιατί βέβαια έχει κάνει πολλή δουλειά και ήταν όλα αυτά πολύ σημαντικά. Το υπόβαθρο το γνωρίζουμε. Για τη μείωση της φτώχειας και την εξασφάλιση της ε, επισητιστικής ασφάλειας, η γεωργία παίζει ένα πρωταρχικό ρόλο. Και αυτή τη στιγμή αυξάνεται η ζήτηση σε γεωργικά προϊόντα και ξέρουμε πως μέχρι το 2050 θα είναι δύσκολο να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χαιρετίζω τις θετικές πτυχές της έκθεσης. Λέει πως θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσουμε τον αναφοδιφασμό των επιστηστικών στους πολίτες Ευρώπης με ε, υψηλά θρεπτικά ε, τρόφιμα. Σημασία λοιπόν της γεωργίας για τον ανεφοδιασμό και την εξασφάλιση του επισητισμού, ε, της Ευρώπης είναι πρωταρχικός. Έχουμε λοιπόν 79%, εκατομμύρια μεσοχτέ Ευρωπαίους που ζουν κάτω από το κατόφλι της φτώχειας και 16%, που, 16 ε, εκατομμύρια που σητίζονται σε συσίτια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει οι γεωργοί να παράγουν και να, να βάζουν τα προϊόντα στην κατανάλωση στην τοπική τους αγορά και θα πρέπει τα τρόφιμα αυτά να είναι θρεπτικά, επαναλαμβάνω. Νομίζω λοιπόν πως για να το πετύχουμε αυτό η ΚΑΠ του μέλλοντος θα πρέπει να δει τι πολιτικές θα προτείνει στον κλάδο αυτό και γίνεται μία αναφορά ε, στους ε, ντόπιου γεωργούς που παράγουν για την ντόπια αγορά. Αυτό θέλουμε να το ενθαρρύνουμε. Το σημείο 28 Μιλάμε για γεωργία μικρής κλίμακας που στέλνει νοπά προϊόντα στις αγορές. Οι μικρές εκμεταλλεύσεις, οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις είναι σημαντικές για την Ευρώπη. Θα πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν αυτή την οικογενειακού τύπου γεωργία, να την προωθήσουμε περισσότερο μέσα στη νέα ΚΑΠ. Χαίρομαι λοιπόν για τα διάφορα συσίτια στα σχολεία, προγράμματα διανομής γάλακτος κτλ. Νομίζω πως ήταν πολύ επιτυχημένα και εξασφαλισμένα επιβάλλησαν πως οι νέοι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν πρόσβαση σε θρεπτική τροφή. Για τους νέους γεωργούς το 2024 στηρίζω αυτή την έκκληση για μέτρα τα οποία θα πρέπει να ισχύσουν για να ενισχυθεί ο ρόλος που παίζουν οι νέοι γεωργοί στον κλάδο. Η συγγήτρια ήδη αναφέρθηκε στο ότι μόνο 7% των γεωργών στην Ευρώπη είναι κάτω από την ηλικία των 35 ετών, ενώ αντίθετα 4,5 εκατομμύρια γεωργοί θα συνταξιωθούν τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη πολύ σοβαρά και νομίζω πως έφτασε η ώρα ενδεχομένως γιατί στην παρούσα οικονομική συγκυρία όπου υποφέρουν διάφορες οικονομίες εγώ βλέπω ότι στη δική μου χώρα έχουμε επιστροφή των νέων προς τη γεωργία ε, και πραγματικά τα κολέγια γεωργικής εκπαίδευσης ή οι γεωπονικές σχολές έχουν γεμίσει από υποψηφίους γιατί ακριβώς η γεωργία γίνεται πια πιο συμφέρουσα. Τώρα για την κοινωνική ατζέντα, ε, νομίζω ότι εδώ το πεδίο εφαρμογής είναι υπερβολικά ευρύ και ίσως είναι και ασαφής η διατύπωση. Είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει κάτι τέτοιο. Μήπως είναι τα κράτη-μέλη πιο αρμόδια. Να το ξαναδούμε. Ανησυχώ για το τι γίνεται με τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων προϊόντων. Αυτή η η εισαγωγή από τρίτες χώρες δημιουργεί εξάρτηση και ίσως αυτή η εξάρτηση είναι υπερβολική. Για την ΚΑΠ και τις αναπτυσσόμενες χώρες το 30 νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας με προτιμιακό καθεστώς από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και ξέρετε πως αυτό είναι θετικό για τους γεωργούς της αναπτυσσόμενες χώρες. Θα έπρεπε ενδεχομένως λοιπόν να εντάξουμε εδώ μια καινούρια πρόταση σχετική ή να αλλάξουμε κάπως το σημείο αυτό τη διατύπωση. Έχουμε και αρκετά μέτρα τα οποία πιστεύω ότι μπορεί να συζητήσουμε είναι η δημιουργία ενός ε, παγκοσμίου συστήματος για τα τρόφιμα. Ξέρουμε πως το 2007 με την επιστημιστική κρίση είχαμε πολλά προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα προσφέρει ασφάλεια ε, σε τέτοιες χρονικές, χρονικές περίοδου επιστημιστικής κρίσης θα εξασφαλίζει τον ανεμφοδιασμό. Θέλω να γίνει η συζήτηση που πρότεινε η συγγήτρα και πιστεύω πως θα πρέπει να εντάξουμε στην έκθεση και κάποιους χώρους στους οποίους αισθανόμαστε κάποιους κλάδους στους οποίους ανησυχούμε ιδιαίτερα. Πάντως σίγουρα θα συνεργαστούμε και νομίζω ότι όλες οι ιδέες θα ακουστούν. Τις καλύτερες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για την έκθεση της ηγήτριας. Ευχαριστώ. Η κυρία Καλνιέτε, παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, γιατί πιστεύω πως η έκθεση αυτή είναι ζωτική σημασίας. Η γνωμοδότηση αυτή υπογραμμίζει το πρόβλημα της ασφάλειας του διατροφικού ανεφοδιασμού και μας δείχνει και ποιες είναι οι στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει έναν, έναν ηγετικό ρόλο για να εξασφαλίσουμε τα αποθέματα τροφίμων. Μόνο η παγκόσμια συνεργασία μπορεί να εξασφαλίσει ε, τη σύντηση του πληθυσμού μας και θα πρέπει η ευρωπαϊκή ασφάλεια των τροφίμων, η ευρωπαϊκή επιστηστική ασφάλεια θα πρέπει να τεθεί στην κορυφή της ατζέντα, γιατί βέβαια η αγορά είναι εξαιρετικά ανήσυχη. Θα πρέπει λοιπόν να μείνουν οι γεωργοί στην Ήπεθρο και να διατηρήσουμε το περιβάλλον εκεί. Ο στόχος αυτός θα, μπορεί να συνδυαστεί, να συνδυαστεί και με μια απελευθέρωση του εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν χρειάζεται λοιπόν εμείς να τοποθετούμε εμπορικά εμπόδια και προσκόμματα σε συναλλαγές όπου δεν χρειάζονται. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν μπορούμε στη νέα ΚΑΠ να συμπεριλάβουμε και κάποιες ε, προτάσεις σχετικές. Πολύ ωραία. Ο κύριος Χάσουορ θα έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια για τις εξαιρετικές της προσπάθειες. Χαίρομαι που αναγνώρισε πως το θέμα της επιστημιστικής ασφάλειας, της τροφικής ασφάλειας θα πρέπει να είναι από τα πιο σημαντικά που αντιμετωπίζουμε. Αυξάνεται συνέχεια ο πληθυσμός της γης. Είναι εξαιρετικά ευμετάβλητες οι τιμές. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό θα αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα, στρατηγική προτεραιότητα για το μέλλον. Ήθελα να τονίσω πως για τις δημοσιονομικές προοπτικές που ακολουθούν περιορισμένο προϋπολογισμό. ΚΑΠ και για τη γεωργία είναι ουσιαστικό να στείλουμε ένα μήνυμα που θα λέει πως η διατροφική ασφάλεια που θα εξασφαλίσει τον ανεφοδιασμό 5 δισεκατομμυρίων πολιτών είναι πολύ σημαντικό και δεν θα πρέπει η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ να περιοριστεί σε κάποια ε, περιφερειακά θέματα για να το πω έτσι. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τρεις απειλές που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Καταρχήν, έχουμε πρόβλημα με την εικόνα που στέλνουμε. Γιατί για πολλούς εδώ στο Κοινοβούλιο τι σημαίνει η ΚΑΠ. Σημαίνει βουνά βουτύρου, λίμνες κρασιού, εικόνες από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Δεν ισχύουν αυτά πλέον σήμερα όμως δυστυχώς αυτές τις εικόνες τις κουβαλάμε μαζί μας και στις διαπραγματεύσεις που πηγαίνουμε και στον τρόπο μας αντιμετωπίζει ο κόσμος. Αυτή είναι η εικόνα μας. Δεύτερον, έχουμε μία αδυναμία στην Ευρώπη και το είπε πολύ σωστά η συγγήτρια, είμαστε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας τροφίμων στον κόσμο. Εισάγουμε 35 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργιών, δηλαδή το μέγεθος της Γερμανίας. Άρα λοιπόν ξέρετε πως εμείς είμαστε πολύτιμη αγορά για πολλούς στον κόσμο σήμερα και φοβάμαι ε, πως σημαίνει το εξή τις διμερείς συμφωνίες που υπογράφονται κάθε στιγμή με το Μερκοσούρ και τα λοιπά, με τον Καναδά και άλλες περιοχές. Η Γεωργία θεωρείται πως αποτελεί το πρόβλημα για τους υπόλοιπους κλάδους. Δηλαδή μπλοκάρουν τα γεωργικά θέματα την επίτευξη συμφωνιών. Και μας λένε, μα κοιτάξτε, θα πρέπει τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα βιομηχανικά ε, ήδη να προωθήσουμε και όχι τα γεωργικά. Όμως, όπως είπε πολύ σωστά η συγγήτρια, τα αποθέματα τροφίμων στον κόσμο αυτή τη στιγμή μειώνονται δραματικά. Εγώ πήγα σε μια διάλεξη χθε το βράδυ που πρόλεψε πως μέχρι το 2050 η Ινδία δεν θα έχει πια νερό μειώνονται τα ενεργειακά αποθέματα. Αυτά θα αποτελέσουν όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα για το μέλλον. Αν λοιπόν αγνοήσουμε τη γεωργία και την ε, ασφάλεια τη διατροφική, την επιστημιστική, τότε θα κινδυνεύσουμε. Ένα τελευταίο. Εδώ έχουμε και κάποια ηθική επιταγή. Ε, εμείς οι αναπτυγμένε χώρε του κόσμου είμαστε Είμαστε εξοικειωμένοι με το γεγονός πως υπάρχει ένα δισεκατομμύριο κόσμου που ζει κάτω από το κατόφλι της φτώχειας στον κόσμο. Θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να παράγουν τρόφιμα για να θρέψουν τους πληθυσμού τους. Γιατί όταν εμείς τα πιο πλούσια κράτη βγαίνουμε στην αγορά και αγοράζουμε τρόφιμα, αυξάνουμε τις τιμές. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ε, σήμερα είναι ένα δισεκατομμύριο και δεν έχουν λεφτά για να φάνε γρήγορα θα γίνουν δύο δισεκατομμύρια. Λοιπόν το μήνυμα είναι πολύ σωστό ε, κυρία μου και νομίζω ότι πρέπει να σας ε, συγχαρούμε για αυτή την επιτυχημένη γνωμοδότηση. Ο Ζωζέ Μποβέ έχει τον λόγο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω. Μόλις έλαβα μια είδηση που ίσως μάθατε κι εσείς. Ο νέος Γενικός Διευθυντής της ε, Διεύθυνσης Γεωργίας ε, από την 1η Ιανουαρίου ε, έχει μεταφέρεται στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Σίλβα Ροδρίγκες Μαγουέλ είναι ο νέος Διευθυντής. Ε, είναι ο παλιός Γενικός Διευθυντής που ήδη έχει ηγηθεί της Γεωργίας. Του εύχομαι κάθε καλή τύχη και δίνω το λόγο στο Ζωζέ Μποβέ. Ε, χαίρομαι να ακούω καλά νέα σε αυτή την αίθουσα, οπότε ε, ευχόμαστε στον κύριο Ντεμαρτή καλό ταξίδι. Ε, νομίζω ότι είναι μια, ένα καλό ξεκίνημα για να αναθεωρηθεί η κοινή γεωργική πολιτική. Ίσως είναι προσωπική μου άποψη την οποία δεν συμμερίζονται όλοι. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή διότι από τις 11 ως τις 17 Οκτωβρίου 2010 έλαβε έλαβε χώρα η πρώτη ε, συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής της Διατροφικής Ασφαλείας από όταν καταρτίστηκε και ναι μεν τα κράτη ψηφίζουν και οι οργανώσεις των ε, γεωργών και των πολιτών συμμετέχουν. Πρέπει λοιπόν σε αυτή την διεθνή διεργασία να ε, περιληφθεί και η εργασία αυτή της ε, ε, εκθέσεως διότι επανατοποθετεί το θέμα εις ε, τη διεθνή σκηνή. Γι' αυτό θύμισα αυτήν την ε, συνεδρίαση η οποία τόνισε τρία στοιχεία που υπάρχουν στην έκθεση και ενισχύει την έκθεση. Καταρχήν το θέμα της κερδοσκοπίας διότι η κερδοσκοπία είναι το βασικό θέμα. Είναι λιγότερα η ε, κερδοσκοπία για κλιματολογικούς λόγους και περισσότερο για λόγους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τις γεωργικές αγορές και υπάρχει μια μετατόπιση της κερδοσκοπίας τώρα από προς τη από τα, τις οικοδομές και άλλους τομείς προς τα γεωργικά προϊόντα. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει στο G20 και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ενισχύσει τη θέση του και να τονίσει σαφώς ότι δεν μπορούμε να κερδοσκοπούμε για τις γεωργικές πρώτες ύλες. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σωστά σε ένα κερδοσκοπικό σύστημα. Το δεύτερο θέμα ήταν η έκθεση που αναφέρεται στις κλιματολογικές αναταραχές και στην ε, ε, υπερθέρμανση της ατμοσφαίρας. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις και να καταπολεμήσουμε τις αιτίες ε, του φαινομένου του θερμοκηπίου. Δεν πρέπει ε, απλούστατα να αναφερθούμε μόνο στη γεωργία αλλά σε όλες τις βιομηχανίες γιατί οι πρακτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται και οι σπατάλοι, οι ενεργειακοί επηρεάζουν τη διατροφική ασφάλεια και πρέπει να το τονίσουμε σαφώς. Τρίτο θέμα το οποίο επίσης ε, ε, έχει απορριφθεί είναι και πρέπει να ενισχυθεί είναι να προστατεύσουμε κοινωνικά τους μικρούς παραγωγούς του, του νοτίου χώρου για να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουν να παραμείνουν στις εκμεταλλεύσεις τους και έχουμε έτσι στο τέταρτο θέμα το οποίο δεν είδα να περιλαμβάνεται στην έκθεση και αναφέρεται εις ε, το land grabbing ε, ε, δηλαδή την υποκλοπή των εκτάσεων. Μπορούμε δηλαδή να δεχθούμε τρίτες χώρες ή επιχειρήσεις να καταλαμβάνουν εκτάσεις σε άλλες χώρες για δικό τους συμφέρον. Είναι αντίθετο και εις τους κανόνες ε, κυριαρχίας των κρατών και τους κανόνες του ΠΟΕ και τώρα είναι ένα ουσιαστικό θέμα το οποίο έχει εξεταστεί στο G20 και θα έπρεπε να εξεταστεί πολύ πιο στεναρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρξει μία ψηφοφορία ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, να τονίσουμε ότι θα πρέπει να εμποδίσουμε την υφαπαγή γεών, το land grabbing για οποιοδήποτε λόγο. Η κυρία Μαγκίνες έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την συνεργασία της και γιατί ενέταξε πολλές από τις ανησυχίες μας σε αυτήν. Ε, θα κρατήσω το λόγο για λίγη ώρα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα και νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί σωστή ισορροπία μεταξύ όλων των συμφερόντων. Καταρχήν, ένα από τα ζητήματα για τα οποία πρέπει να μιλήσουμε είναι το θέμα του πετρελαίου και της γεωργίας και της ενεργειακής συνεισφοράς της ε, γεωργίας όταν μιλάμε για επισητιστική ασφάλεια. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το... είναι κάτι που συνήθως αποφεύγουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ε, χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, τρακτό, τρακτέρ και άλλα μηχανικά μέσα και δεν ξέρω τι εναλλακτικά, εναλλακτικές έχουμε αναφέρθηκε σωστά το ζήτημα του νερού και το πρόβλημα που θα θέσει για την ατζέντα της παγκόσμιας επισητιστικής ασφάλειας. Αν επικεντρωθούμε στην συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να δούμε τι συνέβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε τώρα καθαροί εισαγωγή τροφίμων. Και όπως είπε και ο κύριος Μποβέ, ε, υφαρπάζουμε γέες από άλλες χώρες για να τραφούμε. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτή την έκθεση, γιατί έχει ευρύτερες συνέπειες. Ε, ε, ιδιαίτερες ανησυχίες θα ήθελα να εκφράσω τώρα σε σχέση με την ιδέα των τοπικών τροφίμων. Εγώ δεν συμφωνώ απολύτως με τα σχόλια άλλων συνοδέλφων ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι έχει τη θέση του το θέμα των τοπικών τροφίμων, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί σχετικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν, ξέρω αν μπορούν ο καθένας να, η κάθε χώρα να καλλιεργεί τα δικά της και όλοι να αγοράζουν τα προϊόντα από τον τοπικό τους προμηθευτή. Σε μια έκθεση 31 παραγράφων δεν ξέρω Επίσης, η οργανική γεωργία είναι σημαντική. Είναι μια, ένας ειδικός θύλακας της αγοράς με πολύ πολύ μικρό ποσοστό βέβαια. Πολύ μικρό ποσοστό της τροφής παράγεται βιολογικά, οργανικά. Είναι ένας ιδιαίτερος θύλακας και γι' αυτό υπάρχουν και αντίστοιχες ε, τιμές. Ε, εάν επεκτείνουμε την οργανική γεωργία υπάρχουν συνέπειες για την ποσότητα των τροφίμων που μπορεί να παραχθεί. Υπάρχουν ε, συνέπειες για τη βιοπικιλότητα, για τα ενδιαιτήματα. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερες εκτάσεις. Πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε αυτό και η έκθεση να το συμπεριλάβει. Δεν μπορώ να δεχθώ το γεγονός ότι η οργανική γεωργία είναι η απάντηση σε μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, τα θέματα βιοπικιλότητας ενδιαιτημάτων. Η μεγάλη δυσκολία για τη γεωργία είναι πώς να διατηρήσουμε τα κέρδη της παραγωγικότητάς μας. Ε, στην Ευρώπη έχουμε πάει στην άλλη κατεύθυνση. Πρέπει να παράγουμε περισσότερα από λιγότερα από λιγότερους πόρους. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσει η έκθεση. Μέχρι 40% της παραγωγής μας μπορεί να χαθεί μέσω ε, παρασίτων και ασθενειών και ζυζανίων. Ε, είναι ένα ζήτημα αυτό στον, στον αναπτυγμένο κόσμο. Πρέπει να δούμε πώς η καινοτομία και η έρευνα θα μπορέσουν να βελτιώσουν ε, τα, τις εισρωές στη γεωργία και να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ποσότητα της παραγωγής ε, και, στην, και στους αγρούς και κατά τη μεταφορά και την τελική κατανάλωση. Ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ενισχυθεί η διάσταση της έρευνας και της καινοτομίας σε σχέση με την παγκόσμια επισητιστική ασφάλεια. Δεν νομίζω ότι ο δρόμος προς το μέλλον είναι να είμαστε στραμμένοι προς τα πίσω. Πρέπει να έχουμε στρέψει το βλέμμα μας προς τα εμπρός. Οι άλλοι τομείς που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να ενισχύσουμε είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση και η μεταφορά γνώσεων στους γεωργούς τόσο στον αναπτυγμένο κόσμο όσο και ιδιαίτερο στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αποδέχομαι το βασικό επιχείρημα, αλλά νομίζω ότι αγνοείται η πραγματικότητα της μεταρρύθμισης της γεωργικής πολιτικής. Η επιθυμία μας, η επιθυμία μας είναι να αντικατοπτριστούν στην βασικέ στις βασικές πολιτικές ε, ε, οι γνώσεις μας από το τομέα της γεωργίας. Τε πρόσφατα πολλά χρήματα έχουν βγει από τον αναπτυξιακό προϋπολογισμό και έχουν περάσει στην, ανάπτυξη της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το ποσό αυτό όμως αντί να βαίνει αυξανόμενο, βαίνει μειούμενο. Και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε στον αναπτυσσόμενο κόσμο τη δυνατότητα να αναπτύξει τη γεωργία του με βιώσιμο τρόπο, με εφορικό τρόπο. Και αυτό πρέπει να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Ο κύριος Χάσουορθ μίλησε για τις ηθικές επιταγές και συμφωνώ. Τέλος, για λόγους αφήνειας, ε, ακούμε τη μετάφραση και ο υπάρχουν οι όροι food safety και food security που χρησιμοποιούνται εναλλάξ. Νομίζω ότι η ασφάλεια των τροφίμων από την άποψη της ασφάλειας για την προσωπική μας υγεία, αυτό είναι κάτι το δεδομένο. Αλλά η ασφάλεια των τροφίμων υπό την έννοια της ε, επαρκούς ποσότητας τροφίμων είναι άλλο ζήτημα και δεν πρέπει οι όροι αυτοί να χρησιμοποιούνται ε, ως υποκατάστατο ένας του άλλου. Νομίζω ότι πρέπει να παράξουμε κι και άλλα τρόφιμα χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους και με τρόπο που να μην μειώνει περαιτέρω την απώλεια ενδιαιτημάτων και τη βιοπικιλότητα. Κάτι που δεν έχει θυγεί. Αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους νέους γεωργούς όλους τους γεωργούς να επεκτείνουν την παραγωγή τους. Πρέπει να κερδίζουν κάποια χρήματα αυτοί οι άνθρωποι, να έχουν ένα αξιόπιστο εισόδημα και πρέπει να γίνουν κάποια σχόλια για το γεωργικό εισόδημα, όχι μόνο για τους Ευρωπαίους αγρότες, αλλά γενικά. Πρέπει να αναφέρουμε το ζήτημα της ε, εφοδιαστικής αλυσίδας και της ανησυχίας μας για το ότι επικρατούν άνισες συνθήκες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Νομίζω ότι κάποιο κομμάτι αυτού του εισοδήματος που χάνεται εκεί πρέπει να επιστρέφει στους ε, γεωργούς. Αυτά είναι τα σχόλια που ήθελα να κάνω. Έχω υποβάλει και μερικέ τροπολογίε. Πάντω έχει μεγάλη σημασία να προχωρήσουμε σωστά, γιατί δεν μεταρρυθμίζουμε εδώ μόνο τη δική μα γεωργική πολιτική, αλλά προσπαθούμε να προλάβουμε την εμφάνιση πολύ σοβαρών προβλημάτων που ήδη εντείνονται με την αύξηση του πληθυσμού. Και αυτή είναι μια πελώρια πρόκληση για μα. Ε, θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα με την εισηγήτρια και να υποβάλω μερικέ τροπολογίε. Ευχαριστώ. darf der... Ναι, Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και χαίρομαι που μιλώ μετά την κυρία Μαγκίνες διότι ε, πιστεύω ότι στην έκθεση ε, δεν ε, τονίζει υπερβολικά τις διάφορες πτυχές της γεωργίας αντικατοπτρίζει την κατάσταση πολύ σωστά και εδώ έχουμε την τοποθέτηση της ΦΑΟ ξέρω ότι ζητείτε να αυξήσουμε κατά 70% την παραγωγή και επειδή δεν υπάρχει μία δεύτερη υδρόγειος και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, άλλες μεθόδους πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα γίνει η κατανομή διότι η ε, Ευρώπη και οι Αμερική καταναλώνουν το 50% των τροφίμων ή τα καταστρέφουν δηλαδή υπάρχει τεράστια σπατάλη. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι πρέπει να παράγουμε περισσότερο και όλοι να ζουν όπως ζούμε εμείς. Ε, το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους και αυτό θα αποτελέσει ένα βασικό θέμα για το μέλλον διότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ε, επ' αυτής της οδού και εδώ τίθεται και το θέμα των τεραστίων εισαγωγών διότι έχουμε ένα είδος γεωργίας το οποίο δεν αντικατοπτρίζεται στον υπόλοιπο κόσμο. Ε, η μορφή αυτή η οποία αποτελεί το, το βασικό μας θέμα όταν μιλάμε ε, για σύγχρονη γεωργία ε, εξαρτάται πάρα πολύ από την κατανάλωση ενεργείας και χρησιμοποιεί πολύ ενέργεια. Αυτό είναι πολύ προβληματικό για το μέλλον και γι' αυτό αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν θα μειωθεί το κόστος της ε, ε, ε, γεωργίας ή της ενεργείας αλλά να έχουμε μία γεωργία η οποία θα είναι πιο φιλική στο περιβάλλον, θα χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια και στο μέλλον πρέπει να φροντίσουμε ότι η παραγωγή των βιοκαυσίμων και της βιομάζας να μην υπερβεί τα όρια και να υπάρχει μια ισορροπημένη ανάπτυξη. Το θέμα αυτό ε, θα πρέπει να μας απασχολήσει πιο πολύ διότι πολλές φορές βλέπουμε ότι όταν μιλάμε για τις κλιματολογικές αλλαγές ε, λέγεται ότι πάντοτε πρέπει να μιλάμε για τις κλιματολογικές αλλαγές σε όλες τις εκθέσεις αλλά βλέπουμε ότι πλησιάζει η επόμενη διάσκεψη στο Κανκούν και ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία πραγματικά υπεύθυνη κλιματολογική πολιτική η οποία εξασκείται Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η γεωργία είναι ο, πιο, ο τομέας που πλήττεται περισσότερο και γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε μεθόδους ξέρουμε ε, ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό το χώρο γι' αυτό και είναι ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουμε από κοινού. Τώρα, όσον αφορά τα τρόφιμα και την ασφάλεια, θα σας παραπέμψω ε, στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας που θα παρουσιάσω την έκθεσή μου, όπου θα δείτε ότι υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν ε, πάρα πολύ. Ο, ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Βεβαίως είναι πολύ σωστό ότι εγώ ε, ε, μιλάω τώρα με αυτή τη σειρά διότι ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της έχει πολλά θέματα στα οποία μπορώ να στηρίξω με τους περιορισμούς τους οποίους ήδη έθιξε η σκιώδης εισηγήτριά μας η κυρία Μαγκίνες και θέλω να εκφράσω και άλλη μία ε, κριτική όσον αφορά τις τιμές των σιτηρών όπου ε, αυξήθηκαν 70% ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται ε, με την τιμή των σιτηρών μετά την αύξηση των 70% και βλέπουμε ότι εγώ διαπιστώνω ότι η τιμή ήταν, είναι χαμηλότερη από την τιμή η οποία υπήρχε για τις ζηθοποιίες το 1961 όταν εγώ άρχισα να ασχολούμαι με τον Άρα είναι πολύ χαμηλή και χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρθηκε το σημείο αυτό διότι πρέπει να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε περισσότερους νέους στη γεωργία χωρίς να είμαστε τόσο απεσιόδοξοι διότι διαπιστώνω ότι στη Βαβαρία που είναι μια σημαντική γεωργική ε, περιοχή ή στη Γερμανία έχουμε πάρα πολλούς νέους οι οποίοι ε, είναι έτοιμοι να προσχωρήσουν στο επάγγελμα του γεωργού. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και πιστεύω ότι οι νέοι οι οποίοι παρακολουθούν την κατάσταση ε, ε, ε, είναι, δίδουν μια ευίωνη προοπτική στο χώρο διότι δεν πρέπει να είμαστε πάντοτε απεσιόδοξοι εγώ πιστεύω ότι η γεωργία όπου και να τη συζητήσουμε και σε όποιο χώρο και να αναφέρεται είναι ένας οικονομικός κλάδος ο οποίος έχει πολύ καλύτερες μελλοντικές προοπτικές από οποιοδήποτε άλλος οικονομικός κλάδος είναι κάτι το οποίο πρέπει να το, να τονιστεί και το αναφέρομαι με ε, τέσσερα επιχειρήματα. Πρώτον αυξάνεται ο πληθυσμός της γης και έχει, χρειάζεται περισσότερα τρόφιμα. Δεύτερον δεν θα μπορέσουμε να εμποδίσουμε αν αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο να ε, αλλάξουν και οι διατροφικές συνήθειες διότι στην Κίνα καταναλώνουν κατά μέσο όρο 200 γραμμάρια κρέας την εβδομάδα κάποια στιγμή αντί για 200 θα τρώνε 400 ε, γραμμάρια κατά κεφαλή την εβδομάδα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα χρειαστούμε 13 εκατομμύρια τόνους περισσότερο κρέας και ε, σκεφτείτε τι θα χρειαστούμε ε, σαν αύξηση τροφίμων, τι επίδραση θα έχει στη διαμόρφωση των αγορών και όσον αφορά την ίδρυυση και η ιδίως την ίδρυυση για να μπορούν να ε, χρησιμοποιήσουμε ε, να να πίνουν νερό τα ζώα πόσο χώρο χρειαζόμαστε και δεν αναπτύσσεται σωστά και τέλος θα αυξηθούν οι τιμές ενεργείας θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός και ε, θα πρέπει ε, αν αυξάνεται η τιμή της ενέργειας να πληρώνει ο γεωργός περισσότερα για την ενέργεια που καταναλώνει. Άρα ε, υπάρχει ένας ανταγωνισμός διότι υπάρχουν ορισμένα φυτά ενεργειακά όπως λέγονται που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κακά εδάφη και ε, ε, ε, γιατί να βάζω παραδείγματο χάρη σιτάρι στο χωράφι μου που πληρώνει 1000 ευρώ εάν μπορώ να βάλω φυτά για βιοκαύσιμα τα οποία πληρώνουν 2.500 ευρώ τον τόνο. Άρα η αγορά θα αποφασίσει πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο ανταγωνισμός στο μέλλον. Αυτό όμως που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι θα αυξηθούν πάρα πολύ οι κερδοσκοπίες όσον αφορά τις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Στην έκθεσή μου θα διατυπώσω ορισμένες ιδέες και στην Ευρώπη υπάρχει αυτή η μεγάλη κοινωνία ε, και θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς θα καταπολεμήσουμε την κερδοσκοπία. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν έχουμε ορισμένα ε, θέματα τα οποία να μπορέσουμε να ρίξουμε στην αγορά όταν όταν οι κερδοσκόποι προσπαθούν να ανεβάσουν τις τιμές και νομίζω ότι από πλευράς χρηματοδότησης αυτό δεν πρέπει να είναι προβληματικό ε, διότι ουσιαστικά ε, αν αγοράζει κανείς φθηνά και όλα ακριβά δεν επιβαρύνουμε τον φορολογούμενο και ε, το άλλο που με απασχολεί είναι ο χώρος όπου υπάρχει μεγάλη πείνα. Έχω στενές σχέσεις από ετών με την Αφρική και λυπάμαι αυτούς τους πληθυσμούς διότι οι Αφρικανοί ε, θα μπορούσαν χωρίς μεγάλες δαπάνες να παράγουν ε, τρόφιμα όχι για ένα δισεκατομμύριο άτομα αλλά για δύο. Αλλά δεν υπάρχει σωστή οργάνωση και σήμερα στην Αφρική ε, υπάρχουν ε, άνθρωποι που πεινάνε σε γεωργικές περιοχές βάσει λανθασμένων προγραμματισμών έχω φίλους στην Αφρική και ε, πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την Αφρική και με την πείνα την οποία πρέπει να καταπολεμήσουμε στην Ήπειρο αυτή. Θα ήθελα ε, να πω στην εισηγήτρια και το έκανε και η κυρία Βαγκίνες να καταρτήσουμε μία έκθεση από κοινού διότι η γεωργία στο μέλλον θα έχει πιο μεγάλη στρατηγική σημασία από ό,τι σήμερα πολλοί δεν το έχουν ακόμη καταλάβει και θα πρέπει με αυτή την έκθεση να δείξουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ευχαριστώ. ο κυρίος Κυρέσκη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω δύο λόγια για αυτή τη γνωμοδότηση. Να σας πω καταρχήν πως το θέμα αυτό της επιστηστικής ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό γιατί συζητάμε παράλληλα και τα θέματα του προϋπολογισμού, έχουμε τα θέματα της αναθεώρησης. Θα πρέπει λοιπόν να σταθούμε και να σκεφτούμε με σοβαρότητα το εξής. Πόσα από τα όσα έχουμε πει έχουν ξανακουστεί πολλές φορές στο παρελθόν και κυρίως με ποιο τρόπο αξιολογούμε την ΚΑΠ και τι άποψη έχουν οι υπόλοιποι για την ΚΑΠ. Γιατί μιλάμε τόσο λίγο για τις επιτυχίες της ΚΑΠ. Πώς θα πείσουμε τους πολιτικούς, πώς θα πείσουμε την κοινωνία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε δύο βήματα παρακάτω από τα θέματα τα οποία συνήθως συζητάμε και να προτείνουμε το εξής σε όλα τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό που αφήνουμε, αφήνουμε στην άκρη είναι η λέξη παρεμβατισμός. Την κρύβουμε. Προσπαθούμε να μιλήσουμε για παρεμβατική συμπεριφορά χωρίς να αναφερθούμε στη λέξη αυτή. Εάν όμως δεν έχουμε παρέμβαση, για παράδειγμα, στην αγορά δημητριακών, όπου οι διακυμάνσεις τιμών ουσιαστικά δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Για παράδειγμα, στην εκτροφή πουλερικών, στην εκτροφή χείρων. Εάν λοιπόν δεν παρεμβούμε εμείς, θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους κρίσεις, θα συνεχίσουν οι γεωργοί να κατεβαίνουν στους δρόμους και εμείς τι θα κάνουμε, θα μείνουμε στη γωνιά μας σιωπηλοί χωρίς να βρούμε μία λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε την διακυμάνσεις των τιμών. Δεν μιλάω για παρεμβατισμό όπως είχαμε στο παρελθόν, αλλά στο χώρο, στον κλάδο των Δημητριακών, ε, είναι απαραίτητο να δράσουμε. Τι γίνεται επίσης με το εισόδημα των γεωργών. Μας έχετε παρουσιάσει κάποια στοιχεία για τη συμμετοχή των νέων γεωργών για τους μεγαλύτερης ηλικία, για την κατάσταση των μικρών εκμεταλλεύσεων. Άρα λοιπόν, εξηγήστε μου γιατί δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα πως αυτό που λείπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περισσότερες επενδύσεις στην ΚΑΠ. Δεν θα πρέπει εμείς να θεωρούμε πως η γεωργία μπορεί να αξιολογηθεί μόνο από την οπτική γωνία της επισητιστικής ασφάλειας. Γιατί ξέρουμε ότι και άλλες δραστηριότητες είναι εξίσου σημαντικές για το γεωργικό κλάδο. Όταν μιλάμε λοιπόν για κοινά αγαθά, τι έχουμε στο νου μας, την ενέργεια, τις εκπομπές άνθρακα, τις κλιματολογικές αλλαγές Πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά το νερό, η λειψιδρία, η ξηρασία. Ευτυχώς κάποιος σήμερα το ανέφερε, αλλά ξέρετε πως το νερό θα είναι το βασικό πρόβλημα που δεν θα μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε παραπάνω. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη δημοκρατία, για όλες τις μεγάλες αξίες μιλάμε. Τι γίνεται όμως για να εξασφαλίσουμε την καθημερινότητα των πολιτών μας. Τι γίνεται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για να ξεπεραστούν φυσικές καταστροφές. Τι κάνουμε έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι αυτή που θα βοηθήσει τις υπόλοιπες γωνιές του κόσμου. Νομίζω πως όλα αυτά είναι ιδέες τις οποίες αντιμετωπίζουν πολύ θετικά εκτός Ευρώπης. Δηλαδή, η δική μας παρέμβαση σε δύσκολες καταστάσεις. Είναι πάντα καλοδεχούμενη και βλέπει όλος ο κόσμος που υπάρχει κάποιος που θα τους βοηθήσει, θα τους συντρέξει και βέβαια αυτό βοηθάει και την εντύπωση που έχουν για μας. Άρα λοιπόν με αποθέματα τροφίμων, με υλικό μπορούμε να βοηθήσουμε όσους υποφέρουν. Και τέλος, ας δεχτούμε πώς θα πρέπει με αποτελεσματικό τρόπο να χρησιμοποιήσουμε ε, τους πόρους της ΚΑΠ. Δεν μπορούμε να καταφέρουμε πολλά παραπάνω με λιγότερους πόρους. Μακάρι να μπορούσαμε, αλλά δυστυχώς αυτό είναι ανέφικτο. Θα δώσω τώρα λοιπόν στον επόμενο μιλητή το λόγο. Κυρία Μαγκίνε, σε σχέση με αυτά που είπατε για την οργανική γεωργία, εγώ έχω εξετάσει ε, σε εκτεταμένο βαθμό την, ε, τις οργανικές αρωτρέες καλλιέργειες στην Ανατολική Βρετανία. Υπάρχει η ζώνη πρώτη που είναι σιτηρά, ε, δεν κοστίζει πολύ η παραγωγή του, αλλά αποφέρει πολλά και αυτό είναι καλή επένδυση. Δεύτερη ζώνη, ε, τριφύλι. Ε, η ζώνη αυτή δεν παράγει και πολλά τρόφιμα. Η τρίτη ζώνη, αυτή είναι η ζώνη της καταστροφής. Εκεί έχουν χαθεί εντελώς οι αρωτρές καλλιέργειες, ε, υποφέρουν από ασθένειες, μύκητες κτλ. Ε, εκεί δεν υπάρχει καθόλου κέρδος. Δεν μπορούμε αυτό να το μεταφέρουμε σε μεγάλη έκταση και να πούμε ότι η οργανική γεωργία θα σώσει τον κόσμο. Υπάρχει ρόλος για την οργανική γεωργία, ναι, βοηθάει τη βιοπικιλότητα και ναι, η έρευνα που γίνεται σε ορισμένους τομείς μπορεί να αποβεί πολύ ωφέλιμη κάποια μέρα, αλλά η οργανική γεωργία δεν πρόκειται να θρέψει τον κόσμο. Για την κλιματική αλλαγή τώρα. Νομίζω ότι η Επιτροπή αυτή πρέπει να έχει επίγνωση του από πού προέρχονται όλες αυτές οι ανοησίες. Προέρχονται από το λεγόμενο IPCC, το Διεθνές Κλιμάκιο για την Κλιματική Αλλαγή. Εκείνοι πάλι συνάγουν τις πληροφορίες τους από επιστήμονες που βρίσκονται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Οι, ασθεν... Οι επιστήμονες αυτοί πρώτα έβγαλαν τα συμπεράσματα και μετά ψάχνουν για τα στοιχεία. Ε, Παροτρύνω λοιπόν αυτή την ε, Επιτροπή να διαβάσουμε την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία. Θα δούμε πώς τα άτομα αυτά μοχθούν να περάσουν τη δική τους άποψη και εμποδίσουν τις απόψεις των άλλων να εκφραστούν. Εμείς τα θεωρούμε, τα παίρνουμε, τα παίρνουμε ως γεγονός όλες αυτές τις ανοησίες για την κλιματική αλλαγή και σαν πολιτικοί προσπαθούμε να αντιδράσουμε. Το είδαμε αυτό και πέρυσι με την ε, προσπάθεια διοχέτευσης ε, διοξιδίου ε, του άνθρακα στο έδαφος με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερο τροφή για τα ζώα μας και λιγότερους σπόρους. Τα φυτά σε μια, πλου, σε μια ατμόσφαιρα πιο πλούσια σε διοξίδιο του άνθρακα είναι πιο ανθεκτικά στην ξηρασία. Α, και αυτό είναι πολύ καλό σε σχέση με τη λειψιδρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Ένα παράδειγμα να φέρω. Επανέρχομαι τώρα στο ζήτημα της ε, ξηρασίας και της παραγωγής τροφίμων. Οι πολιτικοί δεν μπορούν να αλλάξουν τον καιρό. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να ενθαρρύνουν τους επιστήμονες να καταστρώσουν σχέδια για τη διαχείριση, την καλύτερη διαχείριση του καιρού. Ονομάζεται βιοτεχνολογία αυτό και πάλι οι γεωργοί τρομάζουν με αυτή την έννοια. Για άλλους πάλι είναι χρήσιμη και υπάρχουν και αντιστάσεις. Και να απαντήσω και στο ζήτημα του νερού. Παρατρύνω την Επιτροπή αυτή να είναι πρακτική, να μην ασχολείται με τα επιφανειακά αυτά θέματα τη οργανικής γεωργίας και κλιματικής αλλαγής, αλλά να δει πώς θα μπορέσει να σημειωθεί πρόοδος. Ευχαριστώ. Κριστόφ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στη Γαλλία έχουμε ένα ρητό. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε που λέει ότι η παιδαγωγική είναι η τέχνη της επαναλήψεως. Δηλαδή να σας πω πόσο είμαστε ε, ειδικοί παιδαγωγικοί εφόσον οι διάφορες παρεμβάσεις επαναλαμβάνουν τα ίδια, τις ίδιες ε, Χαιρετίζω την έκθεση αυτή λοιπόν και τονίζω ότι στη συζήτηση στην οποία βρισκόμαστε το να έχουμε τη δυνατότητα να επαναλάβει το Κοινοβούλιο το βασικό ρόλο της Γεωργίας ε, είναι σωστό διότι για θυμηθείτε πολύ πρόσφατα ε, πώς ε, κοιτούσαμε και πόσο νοσταλγικά κοιτούσαμε τους γεωργούς. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι πολύ βασική η τοποθέτησή μας γιατί δεν θα υπάρχει υπάρχει αλλαγή μόδας όσον αφορά τα ε, ε, τρόφιμα ενώ δεν ξέρουμε για τις εναλλακτικέ λύσεις, ε, ποια θα είναι ε, τα πρότυπα ε, επιβίωσης και πόσο θα εξελιχθούν. Η Γεωργία όμως είναι στρατηγική διότι παράγει αυτό το οποίο οι οικονομολόγοι χαρακτηρίζουν ως ωφέλη για τις περιοχές όπου αναπτύσσονται, δηλαδή πρέπει να δούμε ποιο θα ήταν το δημοσιονομικό κόστος για την Ήπειρό μας αν δεν υπήρχε ε, γεωργία, αν δεν υπήρχε κοινή γεωργική πολιτική και ε, από πλευράς ε, επιδεινώσεως του περιβάλλοντος. Όλα αυτά λοιπόν είναι σκέψεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή. Γι' αυτό εφόσον μιλάμε για ασφάλεια διατροφική και για στρατηγικό χαρακτήρα πρέπει να εστιαστούμε σε τρία θέματα. Τιμές, επίπεδο παραγωγής και όπως το είπα την χρήσιμη γεωργική έκταση και θα επανέλθω στα θέματα αυτά. Καταρχήν για τις τιμές. Εάν ένας τομέας είναι στρατηγικός θα πρέπει οι πολιτικοί ε, να εξετάσουν και να επιλύσουν το πρόβλημα της κερδοσκοπίας. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε ζήσει την οικονομική κρίση, να δούμε πού μας οδήγησαν ε, μας οδήγησε η απουσία ρυθμίσεως και να μην λέμε ότι δεν πρέπει οι άνθρωποι να ε, μην πεινάνε, να ζούνε και να χορταίνουν. Πρέπει λοιπόν ε, να θεωρήσω ότι η διατύπωση της εισηγήτριας είναι ενδιαφέρουσες αλλά δεν νομίζω ότι επαρκούν τα αποθέματα και οι κερδοσκόποι θα ασχοληθούν με το επίπεδο των αποθεμάτων. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει. Βλέπουμε τι γίνεται με το πετρέλαιο, διότι ε, είπατε ε, τι από θέματα υπήρχαν βενζίνης κατά την απεργία για να μην τρέξουν όλοι να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους αλλά ε, δεν πρέπει κανείς να έχει σαν μοναδικό σημείο αναφορά αναφοράς ε, τα αποθέματα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις μετεωρολογικές αλλαγές αλλά επίσης ε, να αποφύγουμε την κερδοσκοπία και να είμαστε τολμηροί. Ε, επίσης θέλω να πω ότι σε μερικά χρόνια η συζήτηση που κάνουμε για το περιβάλλον θα κάνουν τους μελλοντικούς ανθρώπους να χαμογελούν θα πρέπει να βρούμε κάτι πιο περιβαλλοντολογικό γιατί δεν έχουμε επιλογές και δεύτερον εφόσον αυξάνεται ο πληθυσμός της γης και μειώνονται οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις θα πρέπει ή να χρησιμοποιήσουμε καινοτομίε τεχνικές είτε γενικά τροποποιημένους οργανισμούς ή αλλαγές ποικιλιών πιο επιλεγμένες ή ε, επιλογές από πλευράς εκτάσεων συνδυάζοντας διαφορετικά τις παραγωγές αλλά δεν θα, και τις καλλιέργειες αλλά δεν μπορούμε να ε, βασιστούμε σε μία προοπτική μειώσεως της αποδόσεως ένα εκτάριο. Το αντίθετο χρειαζόμαστε και γι' αυτό για να συμφωνήσω με την εισηγήτρια το γεγονός ότι μικρές ε, εκτάσεις μπορεί να είναι πιο αποδοτικές μπορεί να οδηγήσει την κοινή γεωργική πολιτική να πρημοδοτήσει την ενίσχυση για τα πρώτα εκτάρια και όχι τα τελευταία και θα μπορέσει να επιτύχει και μία μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Η σπατάλη και η καταπολέμησή της είναι ε, ηθική επιταγή. Ο καλύτερος τρόπος για να βρούμε νέες ενεργειακές πηγές είναι να μην σπαταλούμε αυτές που ήδη έχουμε. Να σβήνουμε το φως όταν όταν βγαίνουμε από μία αίθουσα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία συγκεκριμένη συμπεριφορά. Εάν όμως συγχρόνως μειώνουμε τη διάρκεια ισχύς των τροφίμων προτού θεωρήσουμε ότι δεν μπορούν πλέον να καταναλωθούν θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε και γι' αυτό συμφωνώ πλήρως με την ιδέα του Ζωζέ Μποβέ ότι δηλαδή πρέπει να γίνει μία συζήτηση ή ένα ψήφισμα για την υφαρπαγή των γεωργικών εκτάσεων διότι ε, είναι σημαντική ε, η γεωργική έκταση αλλά συγχρόνως και ε, η ε, διατροφική ασφάλεια άρα δεν πρέπει να επιτρέψουμε χώρες να χάνουν ε, κυριαρχία σε κάτι που εξασφαλίζει τη διατροφική τους ασφάλεια. Όταν λοιπόν ε, οι μένα αγοράζουν, αγοράζουν εκτάσεις όχι για να παράγουν για την επιτόπια κατανάλωση αλλά για να ξαναπάρουν τα προϊόντα στη δικιά τους χώρα δεν σκεφτόμαστε σωστά και πιστεύω ότι κατά τα άλλα η έκθεση είναι εξαιρετική και μπορούμε να προχωρήσουμε βάσει αυτής. Ευχαριστώ κύριε Μπισού. Και δράτω με τις ευκαιρίες για να θυμίσω σε όλους τους συναδέλφους ότι στις 28 το πρωί αυτή την εβδομάδα, στις 28 Οκτωβρίου, υπάρχει, θα δοθεί μια συνέντευξη τύπου για την Σπατάλη. Και τι κάνει το Κοινοβούλιο πάνω γι' αυτά. Και ο Χέραντς Γκαρσία θα κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ νομίζω θα έθετα επί της ίδιας βάσης ε, με τον κύριο Ντεκού το θέμα αυτό, γιατί όλα όσα είπα αληθεύουν, αλλά υπάρχουν δύο σημεία που είναι πολύ σημαντικά. Καταρχήν, έχουμε το θέμα του επισητιστικού ανεφοδιασμού και έχουμε και τη διατροφική ασφάλεια. Για τον ανεφοδιασμό, ναι, μα αυτός είναι και ο στόχος της ΚΑΠ. Πάντα το επαναλαμβάνουμε. Αρκετά τρόφιμα σε λογικές τιμές για έναν πληθυσμό όπως αυτός της Ευρώπης. Πρέπει να έχουμε επίσης κάποια δίκτυα ασφαλείας, κάποια αποθέματα που μπορούμε να βγάλουμε στην αγορά όταν έχουμε ε, καταστάσεις όπως η αγορά του ε, χειρίου κρέατος Ξέρετε πως η παραγωγή δημητριακών η οποία χρησιμοποιείται για την ε, παραγωγή ζωοτροφών δεν πρέπει να πέφτει στα χέρια κερδοσκόπων. Θα πρέπει λοιπόν οι παραγωγοί να μπορούν κάπου να στραφούν για να αποσμιωθούν κάπου για τις πολύ ψηλές τιμές αυτές. Νομίζω λοιπόν πως αυτή την αγορά ε, Ε, ζωοτροφών και τροφίμων, να παρεμβαίνουμε και εμείς να κάνουμε αποθέματα και να τα διαχειριζόμαστε μετά με τον τρόπο που χρειάζεται. Επίσης, έχουμε, έχουμε πάρα πολλά που έχουμε κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε απογορεύσει πάρα πολλά τα οποία στην, πραγματικότητα δεν κάνουν κακό, αλλά για παράδειγμα ζωοτροφές με ε, ζωικές πρωτεΐνες. Έχουμε πάει αντίθετα στην επιστημονική έρευνα και δεν έχουμε εγκρίνει τη χρήση αυτών των ε, ζωοτροφών, αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους εκτροφείς χείρων ή από τους εκτροφείς πουλερικών. Άρα λοιπόν αυτό που διεκδικούν είναι σωστό. Όπως είπε κάποιος συνάδελφος, αυτή τη στιγμή θα ζήσουμε μια στιγμή απογείωσης απογείωσης της κατανάλωσης πρωτεΐνης, για παράδειγμα, από τον πληθυσμό της Κίνας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήδη αυτή τη στιγμή τρόφιμα τα οποία είναι ακριβά θα διπλασιάσουν και θα τριπλασιάσουν τις τιμές του λόγω αυξημένη ζήτησης. Τώρα για την ποιότητα της, ε, των τροφίμων προσφέρουμε στους πολίτες μας Έχουμε λοιπόν το θέμα της διατροφικής ασφάλειας. Ε, εκεί υπάρχει το θέμα της αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες. Γιατί εάν πρέπει να συνεχίσουμε εξαρτώμενοι από τις αγωγές, γιατί συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις των ΠΟΕ και εξακολουθούμε να δεχόμαστε εισαγωγές, θα πρέπει να τους απαιτήσουμε να σέβονται ένα ελάχιστο κριτήριο ποιοτικό παρόμοιο με αυτό που απαιτούμε από τον κοινοτικό παραγωγό. Εξαιρετική λοιπόν περίπτωση εδώ να υπενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο υπόλοιπο Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Ένωση που θα διαπραγματευτούμε τι τρει δεσμού, ποια είναι η θέση μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε... Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έχουμε περισσότερα ε, με όχι πολύ ψηλέ τιμές και καλής ποιότητας χωρίς να δώσουμε λεφτά στην έρευνα, χρειαζόμαστε μελέτες. Έχουμε να δούμε τι γίνεται με την χρηστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Λοιπόν, πρέπει να δούμε ή πώς θα χρησιμοποιούμε λιγότερους πόρους, ή πώς θα εξορθολογήσουμε τη χρήση των υπάρχοντων, ή πώς τεχνολογικές λύσεις ε, θα μας δώσουν κάποιες απαντήσεις. Δεν μπορούμε να ζήσουμε και άλλη κρίση όπως αυτή με τις τρελές αγελάδες. Ξέρετε ποιο είναι το μέλλον, το βλέπουμε μεσοπρόθεσμα να έρχεται. Γιατί η επόμενη κρίση θα είναι κρίση αξιοποιηστίας του ίδιου μας του συστήματος. Και βέβαια θα πάψουν να μας εμπιστεύονται οι καταναλωτές. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Και για τις ηθικές επιταγές νομίζω ότι τα είπαν οι συνάδελφοι. Θα ήταν απαράδεκτο να μην παρεμβαίνουμε. Και η καλλιέργεια και η εκτροφή ζώων ε, όλη και η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών είναι πολύ σημαντικά. Δεν μπορεί όμως εμείς στην ενέργεια να εξαρτηθούμε από αυτές τις καλλιέργειες από τις οποίες ε, εξαρτώμεθα και διατροφικά. Γιατί καταλαβαίνετε πως αυτό θα μας δέσει τα χέρια στο μέλλον. Έχουμε μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία. Αυτή τη στιγμή αγοράζουν, αγοράζουν εκτάσεις, όχι για παραγωγή, εγώ έχω διαφορετική άποψη. Δεν νομίζω ότι είναι για να παράγουν εκεί τρόφιμα. Όχι. Δεν είναι η γεωργική παραγωγή, η εκτροφή. Όχι. Είναι η εκμετάλλευση των πόρων για, την τεχνολογική, για τον τεχνολογικό κλάδο. Και θα δείτε σε πολλές περιοχές Αφρικής που δεν έχουμε παραγωγή τροφιμών για τον πληθυσμό, αλλά θα είναι για την εξόρυξη, για παράδειγμα, ή την παραγωγή ε, προϊόντων που χρειάζεται η τεχνολογία μας. Άρα θα έχουμε πληθυσμούς που πεθαίνουν και εμείς θα τους παίρνουμε τις εκτάσεις γιατί θέλουμε να αυξήσουμε την παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ε, αυτό είναι απαράδεκτο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Κατρίν Κομπέ. Έχετε τον λόγο. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την έκθεση που ασχολείται με ένα θέμα πραγματικά ουσιαστικό και με πολύ ενδιαφέρον παρακολούθησα όλη τη συζήτηση και τις ιδέες που αναφέρατε. Ξέρετε πως η επισητιστική ασφάλεια είναι μία από τις προτεραιότητες που δίδουμε εμείς και είναι και βασική πρόκληση για την ΚΑΠ τη σημερινή αλλά και την μετά το 2013. Αυτό το οποίο λοιπόν μας ενδιαφέρει εδώ είναι το ότι αποτελεί το σημείο συνάντησης διαφόρων πολιτικών, της γεωργικής, της αναπτυξιακής, αλλά και της εμπορικής και της ενεργειακής, της περιβαλλοντικής, της πολιτικής έρευνας και βεβαίως των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών. Είναι το τέλειο παράδειγμα. Πώς μπορούμε να φανούμε συνεκτικοί μεταξύ αυτών των πολιτικών για να πετύχουμε το στόχο που είναι η επισητιστική ασφάλεια γιατί η συμβολή της ε, ΚΑΠ ε, είναι τεράστια ε, και στην επιστημιστική ασφάλεια αλλά και στην ανάπτυξη. Νομίζω πως κάνει μια πολύ σωστή απογραφή όλων των παραμέτρων η έκθεση. Μιλήσαμε για το θέμα αυτό των εκτάσεων και της υφαρπαγής αυτών των εκτάσεων μιλήσαμε για κάποιες άλλες εμπορικές πρακτικές μιας ανοιχτή εμπορικής πολιτικής γιατί ξέρετε πως όπου εμείς στήσαμε εμπόδια και περιορισμού στο εμπόδιο θυμόσαστε τι συνέβη με την κρίση μετά τώρα πριν από δύο χρόνια μπαίνουμε σε μια ε, βρήκαμε χώρες οι οποίες για παράδειγμα δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του σε ρύζι Άρα λοιπόν αυτό θα έπρεπε να το βάλετε στην έκθεση. Αλλά σε γενικέ γραμμέ συμφωνούμε και τις διαπιστώσεις σας. Και τα αριθμητικά στοιχεία που δίνετε και την ανάγκη που υπάρχει να λάβουμε δράση. Έχω κάποιες παρατηρήσεις για την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ευρω... σε θέματα επιστημιστικής ασφάλειας. Σας υπενθυμίζω τις βασικές δράσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας πω πως υπάρχει το ένα δις ευρώ το οποίο αποφασίστηκε το τέλη του 2008 και αυτή τη στιγμή εκταμιεύεται για την διατροφική κρίση. Η υποχρέωση που αναβάλα που το 2009 στην Λάκυλα στην συνάντηση των G8 είπαμε εκταμίευση 3 δις ευρώ για το 2010-2012 για την, διατροφική ασφάλεια για την επιστημιστική ασφάλεια. Όλα αυτά λοιπόν εμείς θα τα εφαρμόσουμε. Κάτι πολύ σημαντικό, μια σημαντική πτυχή αυτής της πολιτικής είναι η δημοσίευση τον περασμένο Μάρτιο του στρατηγικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά τα επιστημιστικά. Ο κύριος Μποδέ αναφέρθηκε της εργασίας της Παγκόσμιας Επιτροπής Επιστημονικής Ασφάλειας που συναντιέται στη Ρώμη και φαίνεται πως εμείς έχουμε δεσμευτεί και είμαστε πολύ δραστήριοι γιατί σε πολλά διεθνή βήματα είμαστε παρόντες και συζητάμε τα θέματα της επιστημιστικής ασφάλειας. Εμείς, μην νομίζετε, δεν θεωρούμε πως είμαστε ο μοναχικός καβαλάρης, αλλά πιστεύουμε πως πρέπει να συνεργαστούμε με τους διεθνείς ε, εταίρους μας. Δεν θα επιμείνω ιδιαίτερα, αλλά πολύ σημαντικό είναι τα γεωργικά καύσιμα, Σας υπενθυμίζω πως δεν μπορούμε στην Ευρώπη να συσχετίσουμε άμεσα το επίπεδο της καλλιέργειας αυτών των καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται για καύσιμα και της μείωσης της γεωργικής παραγωγής παραδοσιακών τροφίμων, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δύο καύσιμα, χρησιμοποιώντας μόνο 2-3% της παραγωγής δημητριακών. Είμαστε λοιπόν πολύ μακριά από τις αμερικανικές επιδόσεις για τις έντονες διακοιμάσεις των γεωργικών τιμών ξέρετε πως εδώ εμείς έχουμε αναλάβει μια δέσμευση και επίσης την ε, δέσμευση που αναλάβει ο Επίτροπος Γεωργίας για την ε, βελτίωση της διαφάνειας των αγορών ε, πρώτων υλών ψάχνουμε νέα εργαλεία για τη διαχείριση κρίσεων και αυτό αποτελεί ένα σημείο βασικό για τη σκέψη που κάνουμε για την μεταρρύθμιση και αναθεώρηση της ΚΑΠ. Εμείς παρακολουθούμε τις εργασίες της επόμενης G20 και έχουμε συνεργαστεί με τη Γαλλική Προεδρία για να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία. Σήμερα ήδη έχουμε κάποια μέσα στην ΚΑΠ στην διάθεσή μας για να χειριστούμε, για να χειριστούμε τον κίνδυνο, για να εξασφαλίσουμε την ηρεμία στις αγορές και έχουμε επίσης δρομολογήσει και κάποιες πρωτοβουλίες για να βελτιώσουμε τη θέση των γεωργών στην διατροφική αλυσίδα και κυρίως στο γαλακτοκομικό κλάδο. Αυτά είναι κάποια από τα όσα έχουμε κάνει. Βέβαια υπάρχει και μία συνενετική διαπίστωση, μάλλον μια διαπίστωση πως χρειαζόμαστε καινούρια μέτρα. Μιλήσαμε για τα αποθέματα. Δεν είναι εύκολο θέμα. Θυλάκυλα, οι G8 είχαν ζητήσει από τις διάφορους οργανισμούς να δούνε το θέμα αυτό των αποθεμάτων και να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες μας σε πραγματικά και σε θεωρητικά αποθέματα και ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η απάντηση. Δεν έχουμε ακόμα το κλειδί για να εξασφαλίσουμε διαθεσιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξέρουμε και αυτή είναι η εμπειρία μας πως τα αποθέματα είναι πολύ δύσκολα να τα διαχειριστεί κάποιος. Γιατί η σχέση κόστος οφέλους δεν είναι πάντοτε προφανής. Αλλά εκεί που συμφωνούμε είναι πως θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διαφάνεια των αγορών με καλύτερη πληροφόρηση για την παραγωγή, τα αποθέματα, τις τιμές και σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να προωθήσουμε την αποθεματοποίηση σε εθνικό επίπεδο ή σε τοπικό επίπεδο. Και μια τελευταία σκέψη, γιατί στην έκθεση έχουμε μια σειρά στοιχείων για την ΚΑΠ, να σας πω Χρησιμοποιώντας τα σώχη, σε μια προηγούμενη έκθεση η κυρία Μακίνες για την επιστημιστική ασφάλεια, είπε πως η ΚΑΠ θα πρέπει να παραμείνει ακρογωνιαίος λίθος της ευρυστικής ασφάλειας της Ευρώπης και να συνεισφέρει στην παγκόσμια επιστημιστική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο της με δραστήριο τρόπο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και θα ήθελα να σας πω πως έχουμε και διάφορες υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορούν να δώσουν πληροφορίες ή στοιχεία για να εμπλουτίσουν τις συζητήσεις σας. Ευχαριστούμε την Καντρίνα Κομπέτα και τώρα να ξαναδώσουμε το λόγο στην κυρία Σάρμπου. Υπενθυμίζουμε σε όλους τους συναδέλφους ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 8η Νοεμβρίου ώρα 12. Ντατσάνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους συνοδέλφους που έλαβαν το λόγο και που συνέβαλαν με τις ιδέες τους. Ε, σίγουρα θα προσπαθήσω να τα εντάξω όλα αυτά. Ε, αναμένω και τις τροπολογίες που θα υποβάλουν οι συνάδελφοι με μεγάλο ενδιαφέρον. Όλοι συμφωνούμε πάνω σε ορισμένες ε, βασικές ιδέες. Καταρχήν, το θέμα της ρευστότητας τιμών. Δεύτερον, το θέμα των αποθεμάτων, των τροφίμων. Ε, η σημασία της καινούριας ΚΑΠ Υπάρχει διαφορά απόψεων. Υπάρχουν και διαφορές απόψεων ε, στην ε, γεωργία. Από τον τρόπο που το βλέπω εγώ, η βιολογική γεωργία είναι το μέλλον της ε, γεωργίας μικρής κλίμακας. και ας υπάρχουν διαφορές απόψεων για τη βιολογική γεωργία. Τώρα, στο θέμα της διατροφής, η βιολογική γεωργία σημαίνει πιο υγιή διατροφή, πιο υγιεινή διατροφή. Και θέλω πραγματικά να το θέσω στο επίκεντρο όλο αυτό το ζήτημα της οργανικής γεωργίας, γιατί όλες οι μελέτες που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποδεικνύουν προβλήματα με τη διατροφή, με την παχυσαρκία και μια πιθανή, μια δυνατή λύση είναι η ενθάρρυνση του τομέα της οργανικής γεωργίας. Τώρα, για τη στήριξη των νέων γεωργών. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που περιλαμβάνει η έκθεση. Πιστεύω και καταρχήν μιλώ για την εμπειρία της δικής μου χώρας, αλλά νομίζω ότι ισχύει γενικότερα, ότι υπάρχει ανάγκη ενθάρρυνσης ε, των νέων γεωργών και πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, γιατί οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν τη χάνουν σωστής διαχείρισης σήμερα και αυτό οφείλεται στην έλλειψη στήριξης των νέων ανδρών και γυναικών που διαχειρίζονται αυτές τις εκμεταλλεύσεις. Επίσης, έγινε λόγος και για τη γεωργία μικρής κλίμακας και συμφωνώ απολύτως με όσα ελέγχθησαν γι' αυτό. Έγινε λόγος για τη στήριξη της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αλλά αυτό το καλύπτει η έκθεσή μου. Ε, η φαρπογή γεών που αναφέρθηκε από τον κύριο Μποβέ, ε, θα ήθελα πραγματικά να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το θέμα αυτό. Με ανησυχεί όλος εδεωτόρος το ζήτημα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη Γεωργία. Και για το λόγο αυτό το αναφέρω ρητά στην έκθεσή μου. Αλλά μάλλον πρέπει να συμπληρώσω τις πληροφορίες που έχω με πρόσθετα στοιχεία. Κύριε Χάσουουρθ, ναι, συμφωνώ με όσα είπατε, ιδίως για τη σημασία του νερού για τη γεωργία και την ανάπτυξη. Για τις εισαγωγές πρωτεΐνης, ε, πρωτεϊνούχων ε, προϊόντων, δεν, το, δεν ασχολήθηκα εκτεταμένα με το ζήτημα αυτό, γιατί πρόκειται να συζητηθεί. Θεώρησα ότι δεν ήταν ανάγκη να το καλύψω εδώ, δεδομένου ότι δεν θα μπορούσα να τα καλύψω όλα με μια έκθεση. Συμφωνώ με όσο είπε ο κύριος Χαϊσλίχε για τους ε, περιορισμούς στην αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και για το ενεργειακό ισοζύγιο. Γιατί πραγματικά, όπως είπαμε και εδώ, η κλιματική αλλαγή επηρεάζεται καταρχήν από τον βιομηχανικό τομέα και από τον τρόπο με τον οποίο σπαταλούμε τις ενεργειακούς μας πόρους, τους οποίους τους χρησιμοποιούμε ανορθολογικά. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η ρευστότητα των τιμών, η αστάθεια των τιμών. Νομίζω ότι οι τιμές δεν είναι δίκαιες όσο αφορά τους γεωργούς. Υπάρχει όμως μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην τιμή που χρεώνει ο παραγωγός και στην τιμή που αγοράζουμε εμείς το τρόφιμο. Στη χώρα μου ένα κιλό σιταριού ισοδυναμεί με την τιμή ενός καφέ σε μια καφετέρια. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα εύγλωτο παράδειγμα για, την, για το δίκαιο σε εισαγωγικά ε, των τιμών με τους οποίους ανταμείβονται οι εργαζόμενοι στη Γεωργία. Και αυτό ήθελα πραγματικά να το τονίσω όταν είπα στην έκθεσή μου ότι υπάρχει ανάγκη στήριξης από αυτή την άποψη και ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα της ρευστότητας των ε, τιμών, να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Πολλές ιδέες ακούστηκαν ακόμη. Οι περισσότερες είναι πολύ καλές ιδέες. Ε, ασφαλώς δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες αλλά πράγματι ενδιαφέρομαι για τη συζήτηση, για την υποβολή τροπολογιών και θέλω να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη ε, απόφαση που θα συμπεριλαμβάνει όλα όσα εκφράστηκαν εδώ σήμερα και που θα αποτελέσει μια σοβαρή συμβουλή, συμβολή στην συζήτηση που διεξάγεται. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για άλλη μια φορά και όπως είπα Περιμένω με ενδιαφέρον τις έγγραφες προτάσεις και υποδείξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Ε, σου ευχόμαστε καλή συνέχεια, Ντατσιάνα Οκτάβια και φυσικά 8 Νοεμβρίου για την υποβολή τροπολογιών. Ας ολοκληρώσουμε τώρα την συνεδρίασή μας. Οι συντονιστές θα σας ενημερώσουν για τις αποφάσεις που λάβαμε σήμερα το πρωί κατά τη συνάντηση των συντονιστών για τις διάφορες εκθέσεις. Επιπλέον, σας ενημερώνω ότι αποφασίσαμε με τους συντονιστές να υποβάλουμε μια προφορική ερώτηση για το θέμα των ε, ορνήθων, για τις οτόκες όρνηθες. Σας ενημερώνω γι' αυτό και τέλος να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας προγραμματίζεται για τις 15 Νοεμβρίου στις 3 η ώρα. Σας ευχαριστώ. Διακόπτεται η συνεδρίαση της Επιτροπής.